Ladies and Κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε καθίστε. Έχει περάσει το ακαδημαϊκό τέταρτο σχεδόν. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο απογευματινό κομμάτι της συνεδρίασης, αυτή τη φορά από κοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και θα την συμπροεδρεύσουμε με την πρόεδρο Ντανούτα Χίμπνερ, την πρόεδρο της ΑΦΚΟ. Το θέμα αυτού του της διάταξης είναι συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ε, δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για τη δεύτερη εξέταση της έκθεσης ε, που από κοινού έχουν εκπονήσει ο κύριος Μιχαήλ Γκάλερ και ο Εστεμπάν Γκονζάλες Πόνσο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, μετακινήθηκε όχι 10, ήταν 10 Ιανουαρίου, ε, το λέω σωστά έχει περάσει σε κάθε περίπτωση. Οπότε αυτό προς ενημέρωση των μελών και θα ήθελα τώρα να δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Πρόεδρε την Τανούτα Χίμπνερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω επίσης εκ μέρους της Επιτροπής ΑΦΚΟ η προθεσμία έχει παρέλθει για τις τροπολογίες, ε, όπως είπαμε, αλλά αυτή η έκθεση παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέρον ε, μεταξύ των μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε πάνω από 450 τροπολογίες, συνεπώς. Από όσο κατάλαβα, έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά με τη γραμματεία και με τη βοήθεια συμβουλών, ώστε να συντάξουμε τις συμβιβαστικέ και επίσης από όσο κατάλαβα και ελπίζω ότι θα γίνει αυτή τη βδομάδα θα υπάρξει δυνατότητα ε, να υπάρξει συμφωνία επί των συμβιβαστικών ήδη αυτή την εβδομάδα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πρώτα στον Εστεμπάν Γκονζάλες Πόνς και μετά στον Μιχαήλ Γκάλερ. Εστεμπάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους βουλευτές που κατέθεσαν τροπολογίες στην έκθεση. Σίγουρα θα βοηθήσουν οι τροπολογίες, θα διευρύνουν, θα εμπλουτίσουν την έκθεση, θα αποκτήσει μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, ε, γιατί αυτό θέλαμε και ο Μιχαλ Γκάλλερ και εγώ για αυτή την έκθεση, διότι μέρα τη μέρα βλέπουμε να αποκτώλω και μεγαλύτερη βαρύτητα και να γίνεται όλο και πιο επίκαιρη αυτή η έκθεση. Όπως είπε και η πρόεδρος τη Επιτροπής ΑΦΚΟ, 458 συγκεκριμένα τροπολίες κατατέθηκαν. Ε, πήραμε τις μεταφράσεις ε, στις αρχές αυτής της εβδομάδα. Επομένω, ακόμη επεξεργαζόμαστε ενδεχόμενε συμβαστικέ τροπολογίες. Μέχρι στιγμής έχουμε 35 συμβιβαστικέ τροπολογίε, οι οποίε καλύπτουν ένα σημαντικό μέρο ε, των βασικών σημείων τη έκθεση με κάποιε αποχρώσει ε, ε, συμπληρώνουν τις τροπολογίες και ελπίζω ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορέσουμε να δώσουμε στους κοιότητες εισηγητές τις συμβιβαστικές αυτές τροπολογίες για να πάρουμε τις απόψεις τους τουλάχιστον εγγράφος πριν την προηγούμενη, μάλλον πριν την επόμενη συνεδρία που θα έχουμε μαζί τους την 1η Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να σας ε, πω λοιπόν ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η χρηματοδότηση ε, της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όπως ζήτησαν πολλοί βουλευτές. Πάντοτε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διατάξεων από τις συνθήκες και επειδή θέλουμε η Ευρωπαϊκή Άμυνα ε, να έχει περισσότερους οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, θέλουμε να ενισχύσουμε τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευρυμένες εποπτικές ε, εξουσίες για το Κοινοβούλιο, μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτή είναι η στόχη. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα επιχείρηματα της οικονομικής και λιγοτεχνικής αποτελεσματικότητας ε, που δικαιολογούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Συγκεκριμένα θα δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε όθεση στο μηχανισμό ε, δομικής μόνιμης συνεργασίας. Θέλουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ διότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι κάτι στατικό, αλλά θα πρέπει να εξελίσσεται. Ο συνάδελφος Ραμόν Χάουρεγγι το ανέφερε συγκεκριμένα ε, σε μια τροπολογία του. Η νέα γεωπολιτική κατάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη με την απειλή ε, του Ντόναλτ Τραμπ ε, να ε, αποσύρει τη θωράκιση ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΝΑΤΟ. Έχουμε και το μηχανισμό Αθηνά. Θέλουμε να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες, διότι δεν είναι πλέον επιχειρησιακός στην ουσία αυτός ο μηχανισμός. Είναι κάτι που το ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι. Επίσης θα διευρύνουμε τις επεξηγήσεις για τη λευκή βίβλο περί ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε κατόπιν ετήματος πολλών συναδέλφων μια σαφή δήλωση και ορισμό των κινδύνων και των απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να δούμε τι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο και να αναπτύξουμε περισσότερο. Σίγουρα οι τροπολογίε καλύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα, αλλά δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω άλλο. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι υπάρχουν ορισμένες πτυχές ε, που έχουν εισαχθεί μέσω τροπολογιών ε, και τις οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο εδώ στην Επιτροπή. Παραδείγματο χάρη, Ευρωπαϊκός ε, Οργανισμός Πληροφοριών, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό το προτείνει η ομάδα Άλντε. Είναι θετική, φιλόδοξη ιδέα και θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο συντονισμό σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα μέτωπα. Θα θέλαμε επίσης ε, τα κέντρα αριστείας των κρατών μελών ε, να έχουν περισσότερες ε, επαφές. Και η δική μου ομάδα και κάποιοι άλλοι βουλευτές, Ισπανοί βουλευτές από τη σοσιαλιστική ομάδα, ζητούν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου. Και θεωρούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Μέχαλ Γκάλερ προτείνει μια φόρμουλα ώστε στο τέλο τη έκθεση να προσθεθεί ένα προβληματισμό σε σχέση με αυτά που η έκθεση δεν μπορεί να καλύψει, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι τα θέματα προ συζήτηση για το μέλλον. Θα σα πει τα σχετικά νομίζω ο κύριο Γκάλερ. Θεωρώ πάρα πολύ τι προτάσει του. Πολλά άλλα θέματα υπάρχουν που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Το, το σημαντικότερο όμω είναι να ακούσουμε τι δικέ σα θέσει, τα δικά σα επιχείρηματα, ελπίζοντα ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μα με συμβιβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ της κυρίας Προέδρους. Ο ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να θυμίσω κάποια στοιχεία και να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Όντως, στην ε, πολιτική φάση που βρισκόμαστε διαπιστώνουμε συνεχώς αλλαγές τις οποίες δεν τις περιμέναμε κατά ανάγκη σε ό,τι αφορά τι ατλαντικές σχέσει, τώρα έχουμε μια καινούργια κατάσταση, έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία μας αφήνει να καταλάβουμε ότι σε κάθε περίπτωση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών μας θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Βέβαια η ναι, η κυβέρνηση δείχνει έτσι κάποιες ε, τάσεις όχι τόσο φιλικές προς εμάς. Θα πρέπει όμως ε, να αντιδράσουμε και θεσμικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε θεσμικά είναι να βελτιώσουμε αρκετά σημεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τους τομείς αυτούς και να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η συγκεκριμένη συμφωνία έχουμε κάνει λοιπόν, κάποιες προτάσεις τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε στους τομείς αυτούς. Εγώ είμαι της άποψης ότι όντως, όπως είπε και ο συνάδελφος, καταρχάς θα πρέπει όπως λέει και το όνομα, να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορεί να κάνει αυτή η συμφωνία, αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτή τη συμφωνία όταν υπάρχει η πολιτική βούληση. Η δική μου εντύπωση είναι ότι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια η πολιτική βούληση αυξήθηκε για να συνεργαστούμε περισσότερο και αυτά που, προς, που προβλέπει η συμφωνία όπως η μόνιμη ας πούμε, συνεργασία που μπορεί να κινητοποιηθεί ακόμη πιο γρήγορα μπορεί νομίζω να μας οδηγήσει σε ωφέλη για τις κοινέ δραστηριότητες που έχουμε. Ο συνάδελφος ε, ανέφερε και ένα σημείο το οποίο ε, και εγώ έφερα σε συζήτηση σε μια συνάντηση με τους Κιώδης. Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες επί της ουσίας στα θέματα της, ξεπερνούν συγγνώμη, της, τα όσα προβλέπονται από την Λισαβόνα. Νομίζω ότι πρέπει να τις απορρίψουμε γιατί εκπίπτουν και του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας αλλά Ας ε, δούμε καταρχάς δομικά τι θα κάνουμε με αυτές τις ε, τροπολογίες. Ας τις βάλουμε σε ένα τελευταίο κομμάτι ας πούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι όμως για να τις εφαρμόσουμε στα πλαίσια τούτης της συμφωνίας, αλλά για μια μελλοντική συζήτηση πιο γενική που ούτως ή άλλως θέλουμε να κάνουμε για τη συζήτηση και για την ε, συμφωνία αυτή και έχουμε και συμβαστικές προτάσεις και πρέπει να προσέξουμε για ποιες συνθήκες μιλούμε. Γιατί μιλούμε για χρηματοδότηση, Μιλούμε για την κατάσταση όπου οι συνθήκες είναι φυσιολογικές, βρισκόμαστε σε καιρό ειρήνης, αλλά μιλούμε και για περιπτώσεις όπου έχουμε μια αποστολή της ε, GFSP ε, όπου ισχύουν προφανώς άλλοι κανόνες. Καλό είναι λοιπόν να χτενίσουμε λιγάκι τα στοιχεία και να δούμε αυτές τις διαφορετικές νομικές βάσεις πάνω στις οποίες θέλουμε να βασίσουμε τις πολιτικές μας. Αν αυτό το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα. Ας πούμε, όταν μιλούμε για την ε, ε, λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία. Δεν είναι δυνατόν ε, με την ειδική, να, αυτή η πλειοψηφία των κρατών μελών να επιβαρύνει τη χρηματοδότηση για κράτη-μέλη όταν θα ζητήσουμε τη χρηματοδότηση, να περάσει χρηματοδότηση από έγκριση από εθνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε την ειδική πλειοψηφία, η οποία όμως ισχύει για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτά που γίνονται εν καιρό ειρήνη, νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε στα πλαίσια της ειδική πλειοψηφία. Και μια φορά βέβαια μπερδεύονται τα δύο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ακριβεί. δεν ε, δικούμε με ε, ειδική πλειοψηφία σε εθνικό ε, επίπεδο σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν μιλούμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε α, ούτως ή άλλως ισχύει η ειδική πλειοψηφία. Η μόνιμη δομημένη συνεργασία επίσης αναφέρθηκε. δεν είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί προϋποθέσεις για αποστολές σε τρίτες χώρες. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά, αν θέλουν να συμμετάσχουν, να φροντίσουν να συμμετάσχουν όταν θα υπάρξει περίπτωση αποστολή σε τρίτη χώρα. Η ΠΕΣΚΟ δεν σημαίνει ότι θα προετοιμάσει τα πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη να προετοιμάσουν και να παράσχουν τη δική τους συμμετοχή σε τέτοιες περιπτώσει. Αυτό νομίζω ότι δεν ήταν απολύτω σαφές σε κάποιε από τις ε, τροπολογίε που ελήφθησαν. 1η ε, Φεβρουαρίου έχουμε την επόμενη συνάντηση των σκιωδών. Θα λάβετε και σύντομα ε, αύριο κατά πάσα πιθανότητα τις ε, συμβιβαστικές ε, προτάσεις. Μπορείτε να τις δείτε και μετά έχουμε την επόμενη εβδομάδα την άλλη μια δυνατότητα συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι στα πλαίσια του συμβιβασμού νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες πλειοψηφίες και στην ΑΦΕΤ και στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστές, πολύ καλές οι συνθήκες ε, τώρα. Μα ζητείτε να δώσουμε νέες απαντήσεις, γιατί οι παλαιές απαντήσεις δεν αρκούν πλέον για τα ερωτήματα που υπάρχουν. Ούτε για την ε, κατάσταση ασφαλείας της Ένωσης, ούτε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με τους συμμάχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τώρα μια πολύπλοκη διαδικασία να ακολουθήσουμε δίνοντας το λόγο στους Σκιώδης. Η συγητής της ΕΝΤΕ είναι του ΕΛΚ, είναι πρώτη Σκιώδης τώρα η Άννα εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε ε, Στεμπάν Γκονζάλες ε, Πόνσεν και Μακλ για τις προσπάθειές σας. Αναμένουμε με ανυπομονησία τις συμβαστικές ε, τροπολογίες για να δούμε τι διατύπωση προτείνουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει επισημανθεί όταν ε, ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο απόψη ασφαλείας ε, ε, άρχισε να τίθεται υπομφισβήτηση λόγω των δηλώσεων, όχι ακόμα των πράξεων του Πρόεδρου Τραμπ. Είναι λοιπόν ένα κρίσιμο ζήτημα για τα κράτη-μέλη, ώστε να αρχίσουν να σοβαρεύονται όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και να σταματήσουν να παραμελούν αυτό το ύψιστη τη σημασία εργαλείο που έχουν στη διάθεσή του και το οποίο συχνά παραμελούν. Και που συχνά αποτελεί το αντικείμενο διαφόρων ανόητων τσακωμών. Πιστεύω λοιπόν ότι η εκθέση του Κοινοβουλίου μα είναι πολύ σημαντική αυτή τη χρονική στιγμή για να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε όλοι και στο Συμβούλιο ειδικότερα στο θέμα και συμφωνώ. Το σημαντικό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογή της έκθεσης. Το να επαναλάβουμε απλά ότι έχουμε ήδη επαναλάβει πολλά και, σε, ε, και στις εκθέσεις Πάσκου και Μπρόκ θα ήταν ε, περιττό. Και εδώ δεν μιλάμε για το τι υπάρχει μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Μιλάμε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά και αποτελεσματικά το περιεχόμενο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και τα όσα ε, επισημαίνουν οι δύο εισηγητές. Ένας ε, τομέας που μου δημιουργεί πολλές αμφιβολίες είναι το κατά πόσο αρμόζει να μιλάμε για ένα νέο στρατό. Εγώ έχω υπάρξει μέλος της Επιτροπής ε, αυτής από τότε που σχηματίστηκε το 2004. Και κάθε φορά... Το... Και κάθε φορά που μιλάει ο κόσμος ε, για στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερισχύουν ε, όλοι όσοι δεν θέλουν να ενδυναμωθεί η ασφάλεια και η άμυνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας όμως στην ομάδα μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να έχουμε λοιπόν αυτή τον όρο εδώ, εκτός αν πρόκειται για ένα μακροχρόνιο στόχο, που να μην είναι μόνο ε, για το στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ε, ε, ολοκληρωμένες ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον καταστεί απαραίτητο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλά για ένα στρατό, μιλάμε για πολλά περισσότερα. Μιλάμε για όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, για την ασφάλεια και την άμυνα του 21ου αιώνα συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου. Γι' αυτό κατά την άποψή μου είναι προτιμότερο να ασχοληθούμε με το κεντρικά γραφεία της, ε, για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ε, ποιες θα είναι οι σχέσεις, γιατί δεν, μπορεί να υπάρχει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε υπό την προστασία ε, της Δύσης. Αλλά αυτό το είχαμε ήδη αντιληφθεί αρκετοί από εμά τα τελευταία χρόνια, ότι χρειαζόταν επένδυση για την άμυνα και την άμυνα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ότι ήταν σημαντικό να ε, ενισχύσουμε το ρόλο του EDA ε, όσον αφορά τις δημοσίες συμβάσεις, τη διαλειτουργικότητα, ε, τις επενδύσεις στην έρευνα στα διάφορα κράτη-μέλη αλλά και να ενδυναμώσουμε τον εξεταστικό ρόλο αυτού εδώ του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχει μια δημοκρατική εξέταση που μπορεί να γίνει μόνο εδώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το παρόν Κοινοβούλιο όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οποιοδήποτε από αυτούς τους θεσμούς ε, θα παίζει ρόλο στην λήψη αποφάσεων. Οπότε τονίζω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη ενίσχυσης της δικής μας δημοκρατικής εξέτασης και φυσικά έχει να κάνει όλο αυτό και με κονδύλια, με τον προπολογισμό κομμάτι δηλαδή του ευρωπαϊκού προπολογισμού και εκεί πρέπει να είμαστε σαφεί. Σαφώ χρειαζόταν περισσότερο προπολογισμό για την άμυνα των κρατών μελών μας. Αλλά θα πρέπει να προκύψει από επιπλέον κονδύλια ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το σωστό δημοκρατικό έλεγχο και τον ε, ορθό τρόπο χρήση αυτών των κονδυλίων. Είμαι βέβαιη ότι θα έχει τεράστια απόδοση σε σχέση με την επένδυση των χρημάτων των πολιτών μας το να εξετάσουμε σωστά τα πράγματα και αν δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα υπό δημοκρατική εξέταση εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από ό,τι έχουν τα πράγματα στην παρούσα κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη σπαταλούν τεράστια ποσά ε, φόρων των φορολογουμένων για περιττό εξοπλισμό με διπλές εργασίες, ε, με τεράστια παραθυράκια και κενά χωρίς ε, μια σωστή συνεργατική προσπάθεια, όπως απαιτείται απολύτως. Διότι το θέμα δεν είναι να έχει κανείς μόνο τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες, αλλά πρέπει να έχει και το προσωπικό που να έχει εκπαιδευτεί σωστά για τη χρήση τους. Και αυτό απαιτεί περισσότερο από ποτέ συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά ο επαναπροσδιορισμός τώρα και η επέκταση του μηχανισμού Αθήνα ε, που απαιτεί ε, κοινέ επιχειρήσεις να ξεκινήσουν ε, και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλα αυτά. Περιμένουμε υπόμονη λοιπόν, να συνεργαστώ με τους ε, εισηγητέ για το συμβεστικό κείμενο που θα μας παρουσιάσουν. Ευχαριστούμε. Ψάχνω τον Ερή και κυρία Σαμών της ΑΦΚΟ, αλλά δεν τον βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή για να μιλήσει εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ο κ. ο κύριος εκ μέρους του ECR της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη έχω πει την άποψή μου στο Στρασβούργο. Θεωρώ ότι οι αμυντικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να αντίκειται φυσικά ούτε να συγκρούονται με τις υποχρεώσεις μας εναντί του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό που νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε προς το συμφέρον και της Ευρώπης και της παγκόσμιας ασφάλειας θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια καλή, σωστή, λειτουργούσα συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών προσπαθειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σίγουρα δεν θα δεχτώ ποτέ την ε, άποψη του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό είναι το σκεπτικό για τις ε, τροπολογίες που υπέβαλα στο κείμενο των εισηγητών. Επίσης, Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές όταν μιλούμε για τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις των κρατών μέλων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Μόνο ένα μικρό τμήμα των ευρωπαϊκών χωρών πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτό το 2% του ΕΠ δηλαδή, σε επίπεδο δαπανών που απαιτεί το ΝΑΤΟ. Οπότε Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την άμυνα στο επίπεδο που θα καθιστούσε δυνατό να μιλήσουμε σοβαρά για την ανάληψη περισσότερων ευθυνών από την Ευρώπη. Και βεβαίως φυσικά ευχαρίστω θα συνεργαστώ με τους ε, εισηγητές. Ο κύριος Γιώργος Ράντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον ε, κύριο Γκάλερ και τον κύριο Γκονθάλεθ Πόνς για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής και η οποία ελπίζω να συνεχιστεί. Ελπίζω και οι συμβιβαστικέ τροπολογίες ε, που θα ανακύψουν μετά τη συνεργασία μας να είναι ε, οι βέλτιστες δυνατές. Επειδή δεν υπάρχει συνεργασία στον τομέα της άμυνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της δαπανούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς και κανένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό λέει πολλά για την ανάγκη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ορισμένες τροπολογίες που προτείνει η ομάδα Άλντε. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καθήκοντα και υπήρξαν προσδοκίες, τις οποίες δεν έχουμε εκπληρώσει όσον αφορά τυποποίηση στρατιωτικών δυνατοτήτων, αμυντικές αγορές ε, και ούτω καθεξής. Καλούμε λοιπόν με τι τροπολογίε μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση τη κατάσταση. Και καλούμε τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τι δεσμεύσει του, οι οποίε απορρέουν από τα έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίση ε, μια τροπολογία που αφορά τη χρηματοδότηση. Και συγκεκριμένα θέλουμε να συγκριθεί ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε την αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά. για να χρηματοδοτούνται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, με πιο ενιαίο και καλύτερο τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα. Σε ό,τι δεν αφορά κάποιες παρανοήσεις ή την τρέχουσα κατάσταση στις ε, σχέσεις μας ε, με τη ΣΥΠΑ και γενικώ σε σχέσεις, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης ε, για τη Λειτουργία της Ένωσης που μιλάει για συλλογική άμυνα ε, να συμπληρωθεί με συγκεκριμένα μέτρα και τεχνικές για την ενεργοποίησή του, του άνθρωπου αυτού δηλαδή. Και καταλήγουμε και με ορισμένες προτάσεις ε, ίσως πιο ρηξικέλευθες. Για παράδειγμα, αυτή τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών ή Ευρωπαϊκού Στρατού. Βέβαια δεν είναι σαφές κατά πόσο είναι κοινή άμυνα που αναφέρεται, η συλλογική άμυνα ε, που αναφέρεται στο άρθρο που προανέφερα τις συνθήκες, θα περιελάμβανε τέτοια μέτρα ή όχι. Σε ό,τι δεν αφορά την ε, αμυντική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας, περιλαμβάνεται στην έκθεση, πρέπει να περιλαμβάνει πιστεύουμε και αυτή τη διάσταση. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση από αυτού. Πρέπει όμως να ορίσουμε καλύτερα ή τέλος πάντων να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμούς που περιλαμβάνει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης ή άλλα έγγραφα. Ολοκληρώνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κυρίους Πόνς και Γκάλερ και να του ευχαριστήσω εκ των προτέρων και για τις προσπάθειες που θα καταβάλουν να ενσωματώσουν τις ιδέες που προανέφερα στην τελική έκθεση. Αυτό ίσως ως μια προσπάθεια να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά σε μελλοντικά έγγραφα που θα εγκρίνουμε. Για να δούμε αν είναι κανείς από την ΑΦΚΟ κάποιο σκιώδης. Δεν βλέπω κανένα. Ο κύριος Γκέρενς δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι κανείς εκ μέρους του. Ο κύριο Κώστας από την ΚΟΕ. Πασκάλ Ντυρό από τους Πράσινους ή κάποιος εκπροσωπός του. Και μετά Φαβιο Μασίμο Καστάλντο από το EFDD. Όχι. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Υπάρχει και ο Δης ε, της ΣΕΝΤΕ εκ μέρους της ΓΚΟΕ, η κυρία Σαμπίνε Λέζινγκ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Ήδη σε μια προηγούμενη συνεδρίαση είπα στον κύριο Γκάλερ τις βασικές μου παρατηρήσεις ε. οπότε δεν θέλω τώρα να ξαναναφερθώ σε όλα αυτά και το Δεκέμβριο τα είχαμε πει και είχα ξεκαθαρίσει ότι η βασική μας κριτική σε ό,τι αφορά την αυξημένη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το είπαμε και σήμερα και το συζητήσαμε είναι αυτή η καθιέρωση της μόνιμης δομημένης συνεργασίας Πραγματικά ανησυχούμε. Ανησυχούμε με αυτά τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση και σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο. Και ποιες θα είναι οι μελλοντικές αρχές λήψης αποφάσεων για επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, εις οποίες θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν στην ΠΕΣΚΟ κάποιες ε, πτυχές και κάποιοι στόχοι μίλησε ο κύριος Γκάλερ για το ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνουμε τις αρμοδιότητες που μας εκχωρεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να γράψετε τι θέλετε αλλά και τι δεν θέλετε. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Κάποιες φορές έχω την εντύπωση ότι είμαστε πολύ δημιουργικοί και στις λύσεις που προτείνουμε. Και πρέπει να πω ότι αυτές οι λύσεις που προβλέπετε με εντυπωσιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις. Λέτε για φυσιολογικές συνθήκες, εν καιρό ειρήνης. Ότι και υπάρχει ένα επίπεδο. Και πράγματι, αυτές είναι οι συνθήκες και πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένα πράγματα. και μετά λέτε ότι άλλα πρέπει να ισχύουν αν δεν πρόκειται για φυσιολογικές συνθήκες, ε, για την ε, κανονική κατάσταση. Νομίζω ότι συμφωνούμε επί αλλά πρέπει να τηρούμε τις αρχές μας και να εμένουμε στις αρχές ε, των συνθήκων, τις βασικές μας αρχές και τελικά ε, βλέπω ότι είμαι και η μεγάλη υπερασπίστρια της συνθήκης της Λισαβόνας εδώ. Άλλες αρχές για το 2% των στρατιωτικών δαπανών. Το ανέφεραν και οι πράσινοι. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα, από πού θα βρεθούν. Γιατί αν λείπουν αυτοί οι πόροι θα πρέπει να τους πάρουμε από κάπου αλλού. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις για τις εναλλακτικέ που μπορεί να έχουμε. Υποθέτω επίσης ότι στις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες δεν ξέρω κατά πόσον θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ως ομάδα και μάλλον θα καταθέσουμε μια έκθεση μειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δύο συνάδελφοι. Δύο συνάδελφοι είχα ζητήσει. Α, όχι, έχουμε τρίτο. Οπότε να ελέγξουμε λίγο το χρόνο. Ε, ο κ. Φουντσουλίτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Συγχαίρω τους συγητές. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε στο άμεσο μέλλον. Διότι κυρίε και κύριοι, διαμορφώνεται μια νέα τάξη στον κόσμο σήμερα. Δυστυχώς ε, σήμερα παρατηρούμε μια παγκόσμια αταξία ένα παγκόσμιο χάος το οποίο όμως θα λάβει μια νέα μορφή σιγά σιγά θα γίνει μια νέα παγκοσμία τάξη όπου εμείς θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντα των δυτικών χώρων γι' αυτό είμαστε εδώ λαμβάνοντας ε, υπόψη τις 22 χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και η πολιτική άμυνας και ασφάλειας θα διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των συμφερόντων μας στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο είναι απολύτως απαραίτητο να πω ότι ε, για μια φορά συμφωνώ με τα συμπεράσματα ε, των εισηγητών όσον αφορά τη μελλοντική συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επιμείνουμε ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούμε τι δυνατότητε του ΝΑΤΟ σε θέματα ασφαλεία και άμυνα όπω κάναμε και πριν. Τα ε, αρχηγείο του ΝΑΤΟ, του ΣΥΠ χρησιμοποιήθηκε στην ε, στη Βοσνία Ζεγοβίνη όπως θα θυμάστε ε, δεν μπορούμε να σπαταλάμε τα φόρους των φορολογωμένων μας ε, για να χτίσουμε νέα αρχηγεία. Θα χρησιμοποιήσουμε τα αρχηγεία που υπάρχουν ήδη, όπου αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται ήδη. όπου συνάπτονται οι συμφωνίες ε, με τις ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίες και κύριοι, βέβαια, πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ή την ε, κοινή ενωσιακή αμυντική πολιτική, όπως τη βλέπουμε στα κείμενα, αλλά ουδέποτε συζητάμε, ποτέ δεν συζητάμε την κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πυλώνα του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, ε, λέμε τώρα ε, είπατε εκπρόσωπος και, και αντιπρόεδρος και άλλες υψηλές προσωπικότητες στην Ευρώπη λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει δικές της στρατιωτικές και μετικές δυνατότητες διότι κυρίε και κύριοι για να είμαστε μια υπερδύναμη όπως τόνισε η κυρία Μογκερίνη χρειαζόμαστε μέσα χωρίς μέσα και δυνατότητες δεν σε υπολογίζει κανένας Κάθε φορά ε, οι εχθροί σου βλέπουν ένα πράγμα. Τι μέσα, τι δυνατότητες έχεις. Αν δεν τις έχεις τις δυνατότητες, τα υπόλοιπα είναι λόγια χωρίς νόημα. Οπότε για άλλη μια φορά πρέπει να χτίσουμε έναν πυλώνα στο ΝΑΤΟ για την ευρωπαϊκή άμυνα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω να πω στα γρήγορα ότι έχει έρθει η στιγμή της αλήθειας αυτή η έκθεση και ο πρόεδρος Τραμπ μετά όσο έχει πει είναι μια δύσκολη επιλογή ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκό στρατός και είναι σαφές ότι τα όσα έχει πει ο Τραμπ ε, για το ΝΑΤΟ ε, λέει ότι μόνο τα 3,4 ε, κράτη πλέον το 2% του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό το ζήτημα με την Αμερική να πληρώνει το 70% του κόστους του ΝΑΤΟ και να μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Καναδάς μέσα σε όλα αυτά. Είναι μια δύσκολη επιλογή λοιπόν ε, ε, αυτή μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Στρατού και θα χρειαστεί όμως να κάνουμε την επιλογή αυτή. Είτε θα σταματήσουμε τον Ευρωπαϊκό Στρατό και θα πληρώσουμε το 2% για να συμμετάσχουμε στο ΝΑΤΟ, να σταματήσουμε να ε, υπονομεύουμε ή να επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχει ήδη κάνει το ΝΑΤΟ, αποφεύγοντα να δημιουργηθεί ένα υπερκράτο, ή να μην χρηματοδοτήσουμε καθόλου τον Ευρωπαϊκό στρατό και να αφήσουμε το ΝΑΤΟ να διαλυθεί. Και το ερώτημα είναι τι θα καταστήσει την Ευρώπη πιο, ασφαλή. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ του ΝΑΤΟ και θα έλεγα να σταματήσουμε να το υπονομεύουμε. Το δεύτερο, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί υπερκράτος τώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα, ε, ε, δεν είναι ότι είμαστε κάποιο εμπορικό μπλοκ που έχει στρατό. Κανένας δεν έχει τέτοιο στρατό. Οπότε το ερώτημα είναι προς τα που κινούμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα υπερκράτος, έτσι πιστεύω εγώ, ή θα παραμείνουμε ένα εμπορικό, μια εμπορική ομάδα χωρών. Ε, είναι θεμελιώδη σημασία δηλαδή όλο αυτό. Εγώ αντιτίθεμαι προ οποιαδήποτε κίνηση προ, ε, προς όφελο, για τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού στρατού, ευρωπαίων ε, κατασκόπων και με σημαντικέ αυξήσει στον προπολογισμό. Οπότε πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά και να σκεφτούμε τι συνέπειε. Ο κύριο Επιτήδιο, παρακαλώ, από την ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ ε, σύντομο, δεν θα σα απασχολήσω πολύ, διότι το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Η άμυνα και η ασφάλεια είναι δύο πολύ σημαντικές ε, παράμετροι για την ε, ύπαρξη και ενός κράτους και ε, συνασπισμού μιας ενώσεως. Και γι' αυτό πρέπει να το εξετάζουμε με τη δέωσα προσοχή. δυστυχώ. εμείς έχουμε μια ασαφή και όχι ξεκάθαρη θέση για το τι ακριβώς θέλουμε. Μιλάμε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο χρειάζεται να γίνει αυτό και σε τι βαθμό χρειάζεται να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ΝΑΤΟ το οποίο ε, εγγυάται την άμυνα της Ευρώπης και έχουμε και, το, ε, και τις δυνάμεις που συνεισφέρουν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού στρατού οι χώρες προκειμένου αυτός να αναλαμβάνει αποστολές τύπου Πίτερσμπεργκ, δηλαδή ειρηνευτικές αποστολές. Έτσι υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί να διαταράξουμε αυτή την ισορροπία. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε τις ε, αμυντικές ικανότητες ή τις στρατιωτικές ικανότητες ε, μιας ε, χώρας, μιας ενώσεως, θα πρέπει πάνω απ' όλα να καθορίσουμε ποιος είναι ο εχθρός τον οποίο αντιμετωπίζουμε. Μετά να δούμε τι δυνατότητες έχει αυτός ο εχθρός. Και, για να δούμε, και αφού δούμε τι δυνατότητες έχει αυτός ο εχθρός, θα πρέπει να καθορίσουμε μετά τι δυνατότητες πρέπει να αποκτήσουμε εμείς λέμε να δώσουν τα κράτη το 2% από τον προπολογισμό τους. Για να κάνουμε τι. Να αγοράσουμε πόσα όπλα, να κατασκευάσουμε πόσα όπλα. Για να τα στρέψουμε αντίον τίνος. Πώς θα μοιραστούν αυτά τα όπλα. Ποιες δυνάμεις θα τα χρησιμοποιήσουν τα όπλα αυτά. Τι θα γίνουν οι δυνάμεις που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και αυτές που ανήκουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαλυθούν οι μεν και θα ενισχυθούν οι δε. Θα γίνει μια ανάμειξη αυτών. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαφώς το τι θέλουμε και κατόπιν να απαιτούμε από τα κράτη να κάνουν οικονομικές θυσίες. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμία χώρα πλήν της Ελλάδος και της Κύπρου δεν αντιμετωπίζει εξωτερική απειλή. Άρα λοιπόν γιατί να αυξηθούν οι αμυντικές δυνατότητες. Ζούμε σε μια κατάσταση που οι κοινωνίες υποφέρουν, κυρίως στην Ελλάδα με τα μνημόνια υποφέρει ο κόσμος. Πώς λοιπόν θα ζητήσουμε εμείς να δώσουμε τα χρήματα αυτά για να αντιμετωπίσουμε ένα φανταστικό, ένα ανύπαρκτο εχθρό. Ένα εχθρό ο οποίος είναι απλά στη φαντασία μας και όχι στην πραγματικότητα. Αλλιώς ας έχουμε, αν δεν συμβαίνει αυτό που λέω, ας έχουμε την πολιτική ειλικρίνεια και να πούμε ότι αυτός είναι ο εχθρός μας, αυτές οι δυνατότητες έχει, άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να αναπτύξουμε ανάλογες δυνατότητες για να τον αντιμετωπίσουμε. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν έχει νόημα να συζητάμε για αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Thank you very much. And the last speaker... Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ομιλήτρια της ΑΦΚΟ, η κυρία Νταϊάν Τζέιμς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω στη συνεδρίαση. Θέλω να υποστηρίξω τα σχόλια του Βρετανού συναδέλφου μου, του David Campbell Bannerman. Τα είπατε πολύ γρήγορα και εύκολα. Μπράβο, David, είπατε, αναφέρατε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Εγώ ε, συμμετείχα στην εκστρατεία του δημοψηφίσματος, είμαι ευρωσκεπτικίστρια και θέλω να με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, μετά από όσα άκουσα σήμερα το απόγευμα. Η αντιπαράθεση μεταξύ προϋπολογισμού και πόρων. Θέλω και εγώ να επισημάνω ότι ένα από τα θέματα της εξαιρετίας του δημοψηφίσματος ήταν η έλλειψη ε, συμμετοχής από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ και είμαστε έτοιμοι να το πετάξουμε στα σκουπίδια, πού θα βρούμε τα λεφτά, πού θα βρείτε τα λεφτά για να αναπτύξετε τις δικές σας ε, αμυντικές δυνατότητες, χωρίς να πάτε πίσω και να ξαναζητήσετε νέα λεφτά, τα οποία θα έρθουν από πού. Και μετά ήθελα να μιλήσω για το Brexit. Μας αρέσει ή όχι, το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει. είναι ο δεύτερος ή τρίτος οικονομικός συμμετέχων ανάλογα με το πώς το εξετάσουμε και κάποιος θα πρέπει να υπολογίσει με όλα αυτά τα σχέδια, τις ιδέες, ε, όλους αυτούς τους ορισμούς που έχουμε πού θα βρείτε τα λεφτά πρέπει να σκεφτείτε και πώς θα χρηματοδοτήσετε τους πόρους ε, πού θα βρείτε τα λεφτά πρέπει να σκεφτείτε και πώς θα χρηματοδοτήσετε τους πόρους που θα απαιτηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Έλμαρ Μπρόκ. Έλμαρ Μπρόκ. Ich bin immer gerührt <clears throat> über die Europa-Fürsorge der Πάντα συγκινούμε για την ανησυχία που έχουν για την Ευρώπη αυτοί που είναι αντίθετοι με την Ευρώπη, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα δεν είναι πρόβλημά τους πια. Εσείς είπατε το 2019 ότι θα φύγετε, θα είσαστε εκτός με τη δική σας την απόφαση φυσικά. Εγώ λυπούμαι, αλλά ε, τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Για να απαντήσω λίγο στο ποιος είναι ο εχθρό. Στην Σύμβαση της Λισαβόνα λέει ότι υπάρχει αλληλεγγύη των κρατών μελών και σε περιπτώσεις άμυνας. Και επίσης λέει η συνθήκη έμεσα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να έχουμε χώρες που έχουν χαμηλότερα στάνταρ ασφάλειας. Ας πούμε ε, Πολωνία ή χώρες ε, της Βαλτικής. Μπορούμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα έχει το ίδιο επίπεδο και για την ασφάλειά της, για την άμυνά της, όπως και για τους υπόλοιπους τομείς. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι πολίτες μας. Ποιο είναι στα ανατολικά ο εχθρό δεν χρειάζεται να το πούμε, νομίζω είναι προφανέ. Υπάρχουν ε, παραβιάσεις ε, συχνές. Και επίση πρέπει να έχουμε υπόψη μα και το θέμα τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω ένθερμα αυτή την έκθεση που υπέβαλαν οι δύο συνάδελφοι. Ότι όντω δίνουμε πολλά χρήματα. Ο συνάδελφος Γκάλερ νομίζω ήδη το είπε. 200 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται από τα κράτη-μέλη για την άμυνα. 200 δις για την άμυνα δύο φορές τα χρήματα που δίνει η Ρωσία για την άμυνά της. Και έχουμε 1,5 εκατομμύριο α, στρατιώτες. Πάνω δηλαδή, παραπάνω από όσους έχει η Αμερική. Γιατί, γιατί δεν έχουμε κοινή ε, προσέγγιση στη συνεργασία, γιατί ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να έχουμε ένα κοινό, ένα αποθεματικό ανθρωπίνων πόρων και καταλήγουν τελικά τα έξοδα να τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Και τελικά δίνουμε παραπάνω χρήματα και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό το pooling and sharing που είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται, αυτό σημαίνει με τα ίδια λεφτά να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για την εξασφάλιση των πολιτών μας και την ασφάλειά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, αν έχουμε μία περίπτωση όπου Έχουμε συνεργασία Γερμανών Πολωνών ε, ή Γερμανών ε, Ολλανδών και, άλλοι, και άλλες διμερείς ή τριμερείς ε, σχέσεις, όπως για την Europol για παράδειγμα. Μιλούμε δηλαδή για πολυμερείς δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά τους πόρους τους. Και πολλές φορές έχουμε δει να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν επειδή δεν υπάρχει σωστή συνεννόηση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει συνεργασία. Αν μπορέσουμε λοιπόν επιχειρησιακά να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα ή ποιο θα είναι το έξτρα κόστος. Δεν λείπει συνεργασία. Ενίσχυση χρειάζεται αυτής. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν ε, οι νέοι σας εταίροι θα θέλουν να διατηρήσουν το ΝΑΤΟ γιατί λένε ότι είναι και λίγο παροχημένο και λίγο άχρηστο. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών ο νέος, τον είπα. Αλλά δεν βλέπω εδώ με τις δικές μας τις παρεμβάσεις να έχουμε αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Έχουμε ενίσχυση. 80% είναι ουσιαστικά άλλου είδους κόστη έχουμε προεδρικές φρουρέ. και αυτές εντάσσονται μέσα σε αυτά τα πάγια κόστη, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να φτάσουν στο επίπεδο αυτό των δαπανών, του 2% δηλαδή. Αν θέλουμε να έχουμε όμως, θα ήθελα να μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε, αν θέλουμε όντως να εξασφαλίσουμε το ασφαλές μέλλον των πολιτών μας. Και επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση εδώ σε σχέση με αυτά που λέει η έκθεση. Τη ΑΦΕΤ ή άλλες παρόμοιες εκθέσεις που γίνονται, έκθεση που είχα κάνει επίσης και εγώ παρόμοια. Νομίζω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να προχωρήσουν ακριβώς και με βάση των όσων έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι πάντα υπάρχουν συμπεράσματα. Στην εφαρμογή κολλιόμεθα πάντα. Το θέμα είναι η θεωρία να γίνει πράξη. Ελπίζω με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου να μπορέσουμε όντως τη θεωρία να την κάνουμε πράξη. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, I think it was... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ποικίλε διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις για το θέμα αυτό. Η Άννα Γκόμες θα ήθελε το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Ναι, Λυπούμε που ξαναζητώ το λόγο όμως. Ήθελα να απαντήσω στην συνάδελφο James που έκανε αρκετέ αναφορές και σε αυτά που είπα εγώ μεταξύ άλλων. Μιλήσατε για, για το ΝΑΤΟ και είπατε ότι εγώ είπα την είναι Εγώ είπα όχι το αντίθετο, ότι ο Τραμπ ουσιαστικά το ε, στυλιτεύει κατά κάποιο τρόπο και το αχρηστεύει με αυτά που λέει. Και για την ανησυχία που έχετε για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν βάλει την Ευρωπαϊκή Άμυνα ε, χωρί μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, μια από τι χώρε που παρακολεί ε, την ενοποίηση και την ολοκλήρωση τη ε, άμυνα και τη ασφάλεια ήταν η χώρα σα, το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν επιτρέπει και στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό να κάνει τη δουλειά του. Και αν σα ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα χρήματα, δεν πάτε να κοιτάξετε και να μα πείτε τι γίνεται με αυτό το πυρηνικό υποβρύχιο στι ε, ε, αμερικανικέ ακτέ. Κάτι λάθο γίνεται ε, με τα πυρηνικά υποβρύχια που δεν πυροβολούν, που δεν έπρεπε καν να πυροβολούν, αλλά πυροβολούν και προ τη κατεύθυνση. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις πτυχές ασφαλής αμερικανικής πολιτικής μετά την ομιλία του Πρόεδρου Τραμπ για την κατάσταση Τον είπα και έφτασε και ο κύριος Αψαλκάν. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί εξελέγει David Campbell Τέλος πάντων, τα έχω μπερδέψει. Τα έχω μπερδέψει. Ναι, πολύ γρήγορα. Το 2% του ΑΕΠ που είναι ένα 6% ουσιαστικά. Γιατί δεν μπορεί η Γερμανία να το πετύχει για τον Ευρωπαϊκό Στρατό ή τον ΝΑΤΟ. Ό,τι και από τα δύο είναι. Γιατί δεν πετυχαίνει αυτό το 2% η Γερμανία. Η πρόεδρος να ολοκληρώσουμε παρακαλώ εδώ αυτή τη συζήτηση και να εστιάσουμε, αν μου επιτρέπετε παρακαλώ, στην έκθεση. That we have to wrap up. Συγγνώμη, δεν μπορώ ε, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ολοκληρωθεί η γενική συζήτηση και να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας, ε, στον κύριο Γκάλερ και στον κύριο Γκονθάλεθ Πόνς, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Ε, ειδικότερα φέτος ε, η Γερμανία αλλά και πέρυσι αύξησε σημαντικά τον προπολογισμό για την άμυνα. Πρώτον, και η κυβέρνηση των συντηρητικών υπό τον David Cameron στην τελευταία εκστρατεία είπε θέλουμε μείωση στην προεκλογική εκστρατεία την περασμένη φορά. Ο David Cameron ε, έδινε οδηγία να μειωθεί οι αμυντικές δαπάνες. Για τσεκάρατε το κάπου. Αυτό που είπα εγώ είναι να συνεργαστούμε όλοι μαζί ώστε τα χρήματά μας να δαπανώνται αποτελεσματικά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 38 ε, διαφορετικά οχήματα μεταφοράς. είναι γελίο. Κοστίζει ένα σωρό λεφτά. Ο Μάικλ Γκάλερ, τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα κατά τη συζήτηση και θα ήθελα να επαναλάβω για όλους όσοι δεν ε, διάβασαν λεπτόμερο στην έκθεση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ευρωπαϊκό στρατό εντός της έκθεσης. Κάποιες ε, τροπολογίες το αναφέρουν. Ε, και το αναφέρουμε απλά μήπως γίνουν κάποιες συζητήσεις πέραν της συνθήκης ε, για να γίνουν τα πιο σαφή. Δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συνθήκης. Απλά θέλουμε να γνωρίσουμε κάποιες συζητήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Όπως υπόθηκε, ο Πολωνός συνάδελφος ο Ζεσδοφσκή είπε και θέλω να τον καθησυχάσω δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός ούτε σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Απλά πάει πιο πέρα από την υποστήριξη και τη συμπληρωματικότητα. Μιλάμε για καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση των δαπάνων και αυτή είναι μια πρόσκληση προς την ομάδα της ΓΚΟΕ από τη δική σας ε, οπτική γωνία όταν έχετε ερωτήσεις ή επικρίσεις για το 2% γιατί λέτε ότι πρέπει να έρθει από κάπου ναι ξέρετε αν είστε κατά της αύξησης ε, της ποσοστίας αύξησης θα πρέπει να μας δείξετε κάποια δημιουργικότητα για το πώς να βελτιστοποιήσουμε τις δαπάνες οπότε θέλουμε να μας βοηθήσετε να υποστηρίξετε την επιχειρηματολογία για, την καλύτερη, για τις καλύτερες δαπάνες ε, με καλύτερες δημόσιες συμβάσεις, με καλύτερες προμήθειες για να ξεκονομούμε χρήματα για όσους δεν θέλουν να κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια για λίγο παραπάνω δαπάνες τότε να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Δώστε μας καμιά ιδέα. Αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι ότι ενώ εδώ αυτή τη στιγμή ε, συζητάμε για το τι θα γίνει στο μέλλον, ακούω βρετανικές φωνές να λένε «Ναι, σας παρακαλούμε όμως, ό,τι και να αποφασίσετε, φροντίστε όταν εμείς βγούμε φροντίστε να μπορούμε να συμμετέχουμε κάπως στις δραστηριότητές σας. Και χαίρομαι που το ακούω. Ε, ότι φυσικά δεν θέλετε να χτίσουμε τείχους κατά της Βρετανικής συνεργασίας και συμμετοχής ε, αφού θα φύγετε από την Ένωση. Αλλά ακούω και οι βρετανικές φωνές να λένε ότι ε, ε θα είμαστε συνεργατικοί ως εταίροι ε, όταν θα είμαστε εκτός. Έτσι λοιπόν μπορεί να συμμετέχετε περισσότερο από ότι όταν ήσασταν εντός της Ένωσης. Αλλά αυτό από μένα το δούμε. Ε, ευχαριστώ όλους για τις ε, παρατηρήσεις σας. Στις συμβιβαστικές θα τις λάβουμε υπόψη. Ε, κατά την εκπόνηση, ώστε η έκθεση να μπορεί να γίνει αποδεκτή από όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ. Thank you. And now, Gonzalez Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συζήτηση. Συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές συζητά ζητήματα, θέματα που δεν είναι ούτε στις εφημερίδες, ούτε συζητούνται από τον κόσμο στο δρόμο. Σήμερα όμως συζητάμε αυτό που απασχολεί και τους Ευρωπαίους και που το συζητούν. Μιλάμε για ένα θέμα της επικαιρότητα. και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που όταν αυτό το κοινοβούλιο μιλάει για το ενδεχόμενο ευρωπαϊκού στρατού, μιλάει για ένα θέμα της επικαιρότητα, παραλαμβάνω. Πολλές φορές έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Ήταν όμως πάντα θεωρητική. Σήμερα είναι μια πρακτική συζήτηση, διότι έχουν αλλάξει συνθήκες. Ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται αυτό. Αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρουμε τι συνέπειε θα έχει αποχωρησει του. Ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αποσύρονταν από το ΝΑΤΟ ή θα μείωναν τη συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ και θα το κάνουν, θα μειώσουν τη συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα μπορούσαν να είναι σύμμαχο της Ρωσίας. Και σήμερα υπάρχει τέτοιο, και μάλιστα είναι σοβαρό το ενδεχόμενο αυτό, είπα να γίνουν ένα από τους βασικούς συμμάχου της Ρωσία. Χωρί τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη ΣΥΠΑ να δίνουν λιγότερα για το ΝΑΤΟ και να συνεργάζονται ο Πούτιν και ο Ντόναλτ Τραμπ, η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Άμυνας είναι ένα θέμα επίκαιρο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να το αφήσει στη θεωρία. Είναι δυστυχώς πλέον πρακτικό το ζήτημα. Δεν είναι θεωρητικό πια. Η έκθεση δεν είναι στο αντικείμενο το ΝΑΤΟ. Αφήνει εκτός το ΝΑΤΟ. Το θέμα δεν είναι ναι ή όχι ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ ναι, αυτό είναι σαφές. Το θέμα είναι πώς εμείς συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ δεν έχει να κάνει με τον ΝΑΤΟ όμως, αλλά με εμάς, με τη δική μας συμμετοχή στον ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Ενωμένοι ή διαιρεμένοι σε 27 κομμάτια θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η τρομοκρατία τώρα είναι, θα έλεγα, ελάσσον απειλή σε σχέση με μια στρατιωτική απειλή. Όμως η τρομοκρατία μας έδειξε φέτος ότι είμαστε διαιρεμένοι, ότι δεν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση, ούτε τον κατάλληλο συντονισμό και δεν ξέρουμε πώς να οργανωθούμε. Αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, να αντιμετωπίσουμε μια τρομοκρατική απειλή, πολύ λιγότερο ικανοί και έτοιμοι θα είμαστε να, να αντιμετωπίσουμε μια μεγαλύτερη, μια μείζωνα απειλή. Και επίση υπάρχει και το ζήτημα του προπολογισμού. Στα αμυντικά ζητήματα, δύο θέσει μπορεί να έχει κανεί να δαπανά για την άμυνα ή να μην δαπανά για την άμυνα. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρχει είναι το ενδιάμεσο. Δηλαδή να δαπανά για την άμυνα αλλά άχρηστα χρήματα. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 27 αμυντικού προπολογισμού. Και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι 27 αμυντικοί προπολογισμοί σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεται το κόστο αγορά, συντήρηση και επενδύσεων επί 27. Πρέπει να ενωθούν οι προσπάθειες. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πόρων και με λιγότερου πόρου για την άμυνα θα είχαμε πιο πολλά χρήματα για άλλες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μια κοινή προσπάθεια δεν θα μπορέσει κανείς να δαπανίσει περισσότερο. Θα είναι αδύνατον. Θα δαπανούμε όλοι λιγότερο. Αλλά ναι, εάν δαπανούμε 27 κράτη-μέλη τα δικά μας, δαπανούμε 27 φορές παραπάνω. Δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα, είναι πραγματικό το θέμα που συζητούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και ο Μιχαήλ Γκάλερ και εγώ προσωπικά θα κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε οι περισσότεροι κατά το δυνατόν συνάδελφοι να υπερψηφίσουν την έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με τις παρατηρήσεις σας ε, ολοκληρώνεται η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η έγκριση της έκθεσης θα λάβει χώρα στις 9 Φεβρουαρίου στην ΑΦΕΤ και κατά την Ολομέλεια του Μαρτίου στη συνέχεια στο Στρασβουργό. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τα μέλη της ΣΕΝΤΕ παραμείνετε για τα πολύ ενδιαφέροντα επόμενα σημεία της ημερησίας.